δημοκρατία και σε τελευταία ανάλυση περισσότερη ευρώπη. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο την κυρία Γιαννάκου. Ε, κατόπιν του, του ολοκληρώνεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 η ώρα. Περνάμε τώρα στην ε, συζήτηση, για, κοινή συζήτηση ναι, για τέσσερις ε, εκθέσεις. Είναι συζήτηση κοινή για τέσσερις εκθέσεις. Έχουμε λοιπόν ε, τη συζήτηση για τέσσερις εκθέσεις. Θα ξεκινήσει ο κύριος Κάπουλα Σάντος. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η εξωτερική πτυχή της ε, πολιτικής αλίας έχει μια διάσταση πολύ σημαντική. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βασιστούμε στα δικά μας αποθέματα μόνο. Ο κλάδος της Ευρωπαϊκής Αλληλείας αντιπροσωπεύει το 40% μόνο. Το 2009 έχουμε εισαγάγει 15,9 ε, δις ευρώ και εξάγαμε επίσης πάρα πολλά. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Οι διμερείς συμφωνίες με τις τρίτες χώρες είναι σημαντικές. Εάν δεν είχαμε διμερείς συμφωνίες, 3.000 σκάφοι θα είχαν σταματήσει την αλληλευτική τους δραστηριότητα και θα είχαν χαθεί πολλές θέσεις απασχόλησης. Αλλά και οι εταίροι μας έχουν ε, λαμβάνει από αυτές τις συμφωνίες δεν ε, ανταλλάσσουμε μόνο ηχθείες με χρήματα ουσιαστικά. Υπερπροασπιζόμαστε τις δικές μας αξίες. Ενθαρρύνουμε την εφαρμογή και την ιδιοθέτηση των αξιών αυτών και από τους εταίρους μας με τις διμερείς συμφωνίες. Μεριμνούμε για τη διατήρηση των ε, αποθεμάτων και θέλουμε να τηρούνται σωστοί κανόνες ε, στους αλλιευτικούς στόλους. Δηλαδή, η πολιτική αλίας έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει την βιώσιμη και υπεύθυνη αλληλεία και ε, σε περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η εξωτερική διάσταση της πολιτικής αλίας είναι πολύ σημαντική ώστε ο ευρωπαϊκός στόλος να παραμείνει παρόν σε διεθνές επίπεδο και ώστε να υπάρχει παρκής ανεφοδιασμός της ευρωπαϊκής αγοράς. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο καλό είναι να εξετάσει κανείς την έκθεση για την οποία συζητούμε σήμερα ε, με, τη, ε, με τις κομόρες, που έχει να κάνει με τις κομόρες. Δικαίωμα πρόσβασης στα ύδατα των κομορών για 70 ευρωπαϊκά σκάφη με αντιπαροχή, αν θέλετε, χρηματική. συγκεκριμένου ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της αλληλευτικής δραστηριότητας στη χώρα αυτή. Η χώρα αυτή, οι Κομόρες, δεν έχουν άλλους φυσικούς πόρους και μιλούμε ουσιαστικά για τις 33.000 θέσεις απασχόλησης. Προσλαμβάνονται ε, εργασιακό δυναμικό από τις Κομόρες και ε, υπάρχει μέρη ε, ώστε να μην καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ μικρή και έχει δυστυχώς περάσει από διάφορα πραξικοπήματα και έχει μια δύσκολη κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Καλό θα είναι να βελτιωθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας μιλήσω ε, για μια άλλη διάσταση του θέματος και να αναφερθώ και στην έκθεση της κυρίας Γκαλιέ. για να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε σωστά την αλληλευτική δραστηριότητα στις ζώνες 8, 9 και 10 στα ε, πορτογαλικά ύδατα δραστηριότητα που απαγορεύτηκε από 1η Πρώτου του 2010 γιατί ε, τίθενται ε, εν κινδύνο διάφοροι πληθυσμοί ηχθείων χωρίς όμως να υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Γι' αυτό προτείνω να μετατηθεί αυτή η απόφαση για το 2012, ώστε να μπορέσουν οι πορτογαλικές αρχές να εκπονήσουν επιστημονικές μελέτες που να υποστηρίζουν ε, αυτού του είδους ε, το μέτρο. Και είναι μια απόφαση που στηρίζει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Καλό το Κοινοβούλιο να στηρίξει την άποψη αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός 2006 βλέπει την χρηματοδότηση από την κοινή ληφτική πολιτική και το δίκαιο της θάλασσας. Πρόκειται λοιπόν για ένα ε, σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο από κοινού ε, με το Ταμείο της Αλίας είναι ένα από τα δύο βασικά εργαλεία που μπορούμε, μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε κοινή αλληλευτική πολιτική. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες ε, συμπληρωματικές ε, νομοθετικές διατάξεις, τροπολογίες, για να τροπηθεί ο κανονισμός και για να υπάρχει συνέπεια με άλλες νομικές πράξεις. Ε, ε, είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγγύησει ε, και να γίνει προσαρμογή ορισμένων διατάξεων έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες. Πρέπει να διατηρήσουμε τους ε, βασικότερους ε, στόχους και τη δομή που υπάρχει. Διατηρώντας λοιπόν τους ε, στόχους, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι σωστό να υπάρχουν και περαιτέρω τροπολογίες οι οποίες παρότι είναι αρκετά λεπτομερείς μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε όλο αυτό το νομοθετικό έργο να είναι πιο συνεπές με άλλα. Η συζήτηση η οποία έλαβε χώρα πριν και κατά τη διάρκεια της ε, έκθεσης ε, συνέβαλε τα μάλα στη βελτίωσή της η δουλειά της, ε, των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών ήταν πάρα πολύ καλή. Όσον αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση των αληφτικών δραστηριοτήτων, στις τεχνολογίες που υπάρχουν και που επηρεάζουν τον αληφτικό τομέα όπως είναι παραδείγματος χάρη η σύνδεση, η μηχανογράφηση, τα, η μέθοδοι δειγματοληψίας αλλά και η βελτίωση της ποιότητας των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να εισάγουμε μια ε, μέθοδο συγκέντρωσης ε, περιβαλλοντικών δεδομένων, ε, βέβαια και οικονομικών δεδομένων. Να έχουμε τον, ε, την εποπτεία, τον έλεγχο ε, του περιβαλλοντικού τομέα και να ε, διασφαλίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω να σας επισημάνω τρεις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στην έκθεση. Αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο ότι η διαχείριση της αλίας θα πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική γνώση η οποία και αυτή πρέπει να εξυγχρονίζεται. Ε, και αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρείται η βιωσιμότητα αυτής της δραστηριότητας. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συγχρηματοδότησης, του ποσοστού χρηματοδότησης όσον αφορά τη διαχείριση και την χρήση των επιστημονικών δεδομένων και τις ε, πληροφορίες για τα αποθέματα. Το ανώτατο ποσοστό πρέπει να το αυξήσουμε στο 75% Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε τις ε, προνομίες ε, της Επιτροπής. Ε, βεβαίως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν όσον αφορά στην εφαρμογή ελεγκτικών μέτρων στα υδατά τους. Αυτό είναι ένας συμβιβασμός γιατί σας είπα υπάρχει το ανώτατο όριο του 75% ε, και ε, αυτό το αναφέραμε εμείς αλλά και άλλοι συνάδελφοι από άλλες πολιτικές ομάδες που δείχνει λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και τελικά μπορούν να συγκεντρώσουν και την συνένεση στην Ολομέλεια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε συνάδελφε κύριε Φερέρα. Η συνάδελφος Γκρίγε έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, θα αρχίσω την παρέμβασή μου ευχαριστώ τους συναδέλφους για την επικοδομητική τους συνεργασία για αυτή την έκθεση, έκθεση η οποία προκάλεσε ζωηρή συζήτηση. Τόσο, διότι είναι πάρα, πολύ σημαντικ, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι τεχνικές διαδικασίες που διευκολύνουν το έργο των αλλιέων στις περιοχές που ορίζονται από την ε, ε, έκθεση με σκοπό να διαφυλαχθούν τα αποθέματα, στόχους που επιδιώκουν όλοι και συμπεριλαμβανομένων και των αλλιέων. Υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κομισιόν από το 2008 σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτού το μέτρο σε συμφωνία με το Συμβούλιο διότι μόνο αυτά τα δύο θεσμικά όργανα παρέμβαιναν στη διαδικασία. Τα τεχνικά μέτρα ε, διέπονται από ένα παλαιό καθεστώ με τα βατικά μέτρα που διαδοχικά υιοθετήθηκαν, κανονισμό που παρατάθηκε μέχρι το 30 Ιουνίου του 2011, ελήψη συμφωνία με το Συμβούλιο για μια νέα κανονιστική πρόταση που είχε τυπωθεί το 2008 από την Κομισιό με σκοπό την απλούστευση και τη διευκρίνηση τη ισχύουσα νομοθεσία για καλύτερη εφαρμογή των κανόνων και για τη λήψη υπόψη των χαρακτηριστικών δεδομένων Τη Αλία. Τώρα που υπάρχει μια νέα προθεσμία, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Από τη συνθήκη τη Αβώνα, η Αλία υπάγεται σε μεγάλο ποσοστό από τη διαδικασία τη συναπόφαση Το Δικοινοβούλιο έχει λοιπόν αναλάβει το σημαντικό ρόλο του συνομοθέτη που θα ασκήσει προσεγγίζοντα τι απόψει των αλλιέων και των εκπροσώπων τη κοινότητα. Εγώ επειδή ανήκω σε μια θαλάσσια κοινότητα, ε, έχω εκλεγεί σε μια, από μια ε, ε, πόλη που είναι λιμάνι, παρακολουθώ τις εξελίξεις με ιδιαίτερα ενδιαφέρον. ο τομέας της αλίας αντιμετωπίζει κρίση που αυξάνεται. Η σημαντική πρόκληση είναι η αναζήτηση μιας συμφιλίου ανάμεσα στην οικονομική ισορροπία του τομέα και την ε, παροχή ε, ενός εγγυημένου εισοδήματος στους αλίες και την ανανέωση των αλληλευτικών πόρων. Τέλος, το τέλος της εφαρμογής του κανονισμού αρχίζει τη στιγμή που ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την κοινή αλληλευτική πολιτική που θα έχει σημαντικό ρόλο, θα εξασφαλίσει τη συνένεση των αλλιέων, των καταναλωτών και των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα που θα καθορίζουν το ύψος των ποσοστώσεων και την όλη λειτουργία του τομέα. Αυτό προποθέτει ότι θα έχουμε μια ουσιαστική πρόταση της ε, Κομισιόν για την αξέλιξη των τεχνικών μέτρων, κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Μια νέα πρόταση θα πρέπει να μεριμνήσει για την προσαρμογή των τεχνικών δυνατοτήτων και μέσων σε αυτά που ισχύουν στην πράξη, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενου αναζητώντα μια ε, επικαιροποίηση του κανονισμού και με σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Εν ώψη αυτών των προοπτικών, η πρότασή μου είναι να δεχθούμε την πρόταση της Κομισιόν για μια παράταση μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, χωρίς ουσιαστική μεταβολή των τεχνικών μέτρων που ισχύουν αυτή τη στιγμή, με μόνη διαφορά την ε, μάτι δικτυού που χρησιμοποιείται για το βασιλάκι. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ανησυχίες μεταξύ των αλλιέων και των επαγγελματιών. Γι' αυτό υποβάλλω ένα διπλό αίτημα να, να μην υπάρξει, προσαρμογή των τεχνικών μέτρων που ισχύουν αυτή τη στιγμή και, τη... και το ξεκίνημα μιας διαδικασίας διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους εν ώψη του επόμενου κανονισμού. Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να κατατεθεί σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο ώστε να είναι έτοιμος για το 2013. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε άμεσα να δουλεύουμε πάνω σε αυτό τον κανονισμό δεν μπορούμε να προβλέψουμε περαιτέρω παράταση πέρα των 18 μηνών αυτού του κανονισμού. Μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για μια μεταβατική περίοδο. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Θέλω να σας πω ότι οι διερμηνείς πραγματικά είχαν εκπληκτική απόδοση και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Φράγκα. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να αναφέρω τις ε, επιπλοκές που έχουν σημειωθεί με το φάκελο αυτό, διότι και η Επιτροπή και το Συμβούλιο αρνούνται τη ε, δυνατότητα της συναπόφασης που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Γρυλανδία θα πρέπει να εξάγει με τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ωφελεί και τη Γρυλανδία που εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το 80% των αλλιευμάτων της, ωφελεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Δανία, η οποία λαμβάνει κατά κύριο λόγο τις εξαγωγές αυτές. Και μία από τις προϋποθέσεις ε, είναι να δεχθεί η Γρυλανδία τις, ε, τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε θέματα υγιεινής και ε, ε, προστασίας για να μην υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της βασιζόμενη στο άρθρο 203 της Συνθήκης. Δηλαδή, αυτό σήμαινε ότι εμείς απλά μόνο θα μας ζητεί το υγνώμη γνώμη στο Κοινοβούλιο. Η νομική υπηρεσία ε, παρατήρησε την ανομολία αυτή εξ αρχής. Πέρα από το περιεχόμενο και πέρα από το διακύβευμα και τη σημασία που είχε όλο αυτό το θέμα για τη ε, γριλαδία, δεχθήκαμε να συμμετάχουμε σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Τη στιγμή λοιπόν που ε, ήρθε προς ψήφιση, το Συμβούλιο ξαφνικά υιοθέτησε τελείως διαφορετική πρόταση με διάφορες τροποποιήσεις που θέλουν να κρύψουν την προφανή σύνδεση με την κοινή οργάνωση αγορά. και ουσιαστικά έκαναν τη συναπόφαση ένα χειρισμό ανέξοδο. Γιατί ούτω ή το Κοινοβούλιο θα είχε εγκρίνει το κείμενο χωρίς κανένα πρόβλημα. Ε, κληθήκαμε λοιπόν να συζητήσουμε ένα νέο κείμενο και Σαφές ήταν ότι το Συμβούλιο ήθελε να αφαιρέσει ουσιαστικά την εξουσία από το Κοινοβούλιο και γι' αυτό επισήμως ζητήσαμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στην γνωμοδότησή της παραθέτω και λέω ότι είπε το εξής «Στόχος είναι να απαιτηθεί από τη Γρυλανδία να υιοθετήσει τους κοινοτικού κανόνες σε θέματα υγειονομικά ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων στην εσωτερική αγορά και την ε, συμμετοχή της στην ενιαία αγορά όπως, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο» και θα πρέπει η Γρυλανδία να εφαρμόσει τους αντίστοιχους κανόνες που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφάλειας τροφίμων και θέματα υγειονομικά ε, στα αλλιευτικά προϊόντα που εξάγει. Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων γνωμοδότησε ομοφόνος ότι τα άρθρα 203 και 42,3 ε, της συνθήκης αλλά και το πρωτόκολλο 34 το σχετικό για τα προϊόντα που υπόκεινται σε κοινή οργάνωση αγοράς στη Γρυλανδία είναι, ε, συνιστούν τη νομική βάση της πρότασης αυτής. Ως εκ τούτου, ως εισηγήτρια κατήρτισα νέο σχέδιο έκθεσης, τροποποιώντας τη νομική βάση. Και αυτό είναι αυτό που αύριο θα παρουσιάσουμε για να το εγκρίνετε. Και θεωρούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι η πρώτη ανάγνωση αυτή το μόνο που μου μένει να ζητήσω από την Επιτροπή και το Συμβούλιο που νομίζω ότι απουσιάζει από αυτή την αίθουσα να δράξουν αυτή την ευκαιρία για να αναγνωρίσουν τη νέα νομική βάση και να θεωρήσουν και αυτά τα θεσμικά όργανα ε, ότι αύριο γίνεται πρώτη ανάγνωση. Το θέμα δεν έχει να κάνει, το πρόβλημα δεν είναι το περιεχόμενο, το θέμα είναι για τη νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Δαμανάκη ε, εκ μέρους ε, τη επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ηγητές για τις προσπάθειές τους και θα αναφερθώ τώρα κύριε Πρόεδρε μου το επιτρέπετε στην κάθε μια από τις εκθέσει η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης ε, της Κομόρας. Ευχαριστώ τον κύριο Καπούλη Σάντος για, το έργο, για τις προσπάθειές του ως και με χαρά διαπιστώνω ότι η Επιτροπή Ελίας έχει υποστηρίξει θερμά την πρότασή του. Πώς γνωρίζετε, η δέσμευση είναι να προωθούμε και να ενισχύουμε τη βιώσιμη αλία στα ύδατα των εταίρων μας συμπεριλαμβανομένε και της περιοχής του Ινδικού ωκεανού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούν οι διμερείς σχέσεις με τις χώρες αυτής της περιοχής και τις κομόρες ειδικότερα σε σχέση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις, οργανώσεις, στις περιφερειακές οργανώσεις αλίες όπως είναι η οργάνωση για τον τόνο, για την αλία του τόνου. Γι' αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συμφωνία. Σήμερα έχουμε τέσσερις συμφωνίες σύμπραξης στον ειδικό κενό. Σε Ιχέλες, Ματαγασκάρι, Μοζαμβίκη και Κομόρες. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια να υπάρξει με τους Κομόρες μία συμφωνία επειδή η συμφωνία αυτή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για την παρουσία του στόλου μας στην περιοχή αυτή. Επίσης είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το διάλογο στον τομέα των τομεακών πολιτικών για να προωθήσουμε την εφαρμογή μιας υπεύθυνης πολιτικής ελίας σε αυτή την περιοχή. Τώρα θα ήθελα να πω λίγα λόγια, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με το αίτημα του εισηγητή στην Επιτροπή όταν ολοκλήρωσε την έκθεσή του. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να ενημερώνει σταθερά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων πριν από την υπογραφή διεθνών συμφωνιών. Το εννοούμε αυτό ειλικρινά. Θέλουμε να είναι διαθέσιμα όλα τα υπάρχοντα στοιχεία αλλά βεβαίως πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί στη Συμφωνία Πλαίσιο. Στην πράξη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν ε, τηρούν, έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους διαβιβάζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις ίδιες πληροφορίες που διαβιβάζουν στο Συμβούλιο και την ίδια στιγμή. Επίσης, ε, θα σας, δώσουμε την, ε, θα σας υποβάλουμε την αξιολόγηση post και ante των συμφωνιών μας το ταχύτερο δυνατό και αύριο στην ψηφοφορία για την, για την συμφωνία σύμβραξης με τη Μαυριτανία οι περιοχές επιτροπής έχουν φροντίσει ώστε το κείμενο να είναι διαθέσιμο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν αφού ενημερωθούν πλήρως τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μελών του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών σε διεθνείς συναντήσεις, πρέπει να τονίσω ότι η Συμφωνία Πλαίσιο ε, ισχύει για πολυμερείς ε, διεθνείς διασκέψεις. Επίσης, σκοπεύουμε ε, να προωθούμε πρακτικές συμμετοχής σε διμερείς διαπραγματεύσεις. Οποιαδήποτε απόφαση να περιληφθούν ως παρατηρητές τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αντιπροσωπείες λαμβάνεται από το Σώμα των Επιτρόπων κατά περίπτωση μετά από αξιολόγηση των νομικών, διπλωματικών και τεχνικών δυνατοτήτων που αναφέρονται στις συμφωνίες πλαίσια. Αυτό που θα ήθελα να εδώ είναι ότι η στάση των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι πάρα πολύ θετικές. Καταβάλουν κάθε προσπάθεια, καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολυνθεί η συμμετοχή σας. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη έκθεση για τα κοινοτικά μέτρα για την εφαρμογή της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ευχαριστώ την Αρμόδια Επιτροπή και τον ε, εισηγητή τον κύριο Φερέρα για την έκθεσή του. Χάρη στις προσπάθειές τους έχουμε ένα κείμενο μπροστά μας το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο. Με τα χαρά σας λέω ότι το κείμενο αυτό είναι επίσης αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε θαυμάσια συνεργασία λοιπόν ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα για αυτή την υπόθεση και μετά από επιτυχή άτυπη, τρίλογο ή τριμερή διάλογο καταλήξαμε σε συμπεράσματα και θα ακολουθήσει η πρώτη ανάγνωση που θα ε, ολοκληρωθεί επιτυχώς. Η πρόταση αυτή αποτελεί ένα εξορθολογισμό του κανονισμού για το δεύτερο χρηματοδοτικό μέσο, όπως ονομάζεται, που καλύπτει ε, τη... θέματα διακυβέρνησης, συγκέντρωση στοιχείων, επιστημονικών πληροφοριών, και επίσης θέματα ελέγχου και εφαρμογής. Η αναθεώρηση έχει σκοπό να εξασφαλίσει συνοχή, συνέπεια ανάμεσα στο κανονισμό αυτό και άλλα νομοθετικά κείμενα, προβαίνει σε νομικές προσαρμογές και διευκρινήσεις των διατάξεων. Καλό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σχετική πρόταση. Τώρα θα έρθω στην τρίτη έκθεση για τα μεταβατικά τεχνικά μέτρα για τα οποία ευχαριστώ την κυρία Γκρελιέ, την εισηγήτρια. Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να επεκταθούν τα μεταβατικά τεχνικά μέτρα μέχρι το τέλος του 2012. Αυτά βασίζονται στην ε, παραδοχή ότι η ε, μεταβληθήσα, η ε, κοινή αλληλευτική πολιτική που θα έχει μετατραπεί θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του επόμενου έτους και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Η δική μου λοιπόν η πρόθεση προτείνοντας αυτή την παράταση είναι να αποφύγουμε να υπάρξουν περίπλοκες συζητήσεις για τεχνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης. Η Κομισιόν συμφωνεί με αυτά που είπε που ελέγχθηκαν ε, σχετικά με το bore fish ε, επειδή αυτά βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες. Επίσης ε, όσον αφορά το βασιλάκι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που κατέθεσαν επιπρόσθετες τροπολογίες. Ε, οι τροπολογίες αυτές όμως δεν γίνονται δεκτές γιατί δεν έχουν εγκριθεί από τους επιστήμονες ή διότι οι επιστήμονες δεν έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τα κράτη-μέλη για να προβούν σε σωστή αξιολόγηση. Και τέλος επιτρέψτε μου να πω και λίγα λόγια για την έκθεση που αφορά στην εισαγωγή προϊόντων αλίας από τη Γρυλανδία. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής Αλίας, την κυρία Φράγκα, για τη δουλειά δουλειά Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή αφορούν ένα μακροχρόνιο αίτημα της ε, Γρυλανδίας. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο να πλουστεύσουν τα ε, μέτρα τα υγειονομικά, τις διαδικασίες πιστοποίησης και η Γρυλανδία να καταστεί μέλος της κοινή αγοράς για τα προϊόντα λίας και τα υποπροϊόντα τους. Και αυτό ε, συμφωνία απόλυτα με τη συμφωνία του 2006 όπου προβλέπεται να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της Γρυλανδίας και να συνεργαστούμε συνεργαστούμε στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων. Η Κομισιόν με χαρά διαπιστώνει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο ομόφωνα, η Γρυλανδία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών, όλοι λοιπόν είναι πρόθυμοι να τηρήσουν αυτή την υπόσχεση και να υποβάλουν σχετική πρόταση. Και επιτρέψτε μου να καταστήσω σαφές ότι για μας, για την Επιτροπή, η σχέση με τη Γρυλανδία είναι κέρια σημασίας και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε γιατί. Είναι πολιτική προτεραιότητα η Γρυλανδία. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι οι συζητήσεις για τη νομική βάση πάνω στην οποία θα βασιστεί η πρόταση δεν θα θέσουν σε κίνδυνο αυτά τα τόσο σημαντικά μέτρα. Κατανοώ πολύ καλά τις ανησυχίες της κυρίας Φράγκα για τη νομική βάση αυτής της πρότασης και για τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκείνο μπορώ να πω είναι ότι η Επιτροπή δεν θα ε, προκαλέσει κολλήματα στην αναζήτηση ρεαλιστικής λύσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι η νομική βάση της πρότασής μας είναι σωστή, αλλά παρόλα αυτά δεχόμαστε και το διευκρινίζω αυτό ε, αν τελικά ε, το, Συμβούλιο εγκρίνει την άποψη του Κοινοβουλίου, εμείς θα το δεχτούμε. Το Συμβούλιο λοιπόν πρέπει τώρα να ελέγξει τις δυνατότητες που υπάρχουν και να προχωρήσει σε συμφωνία με την ε, συνθήκη. Ελπίζω το θέμα να λυθεί ταχύτατα έτσι ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στις σχέσεις μας με τη Γρυλανδία. Γιατί αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να σας πω ότι επιθυμώ να διευκολύνω κλείνω τη δουλειά της ε, κυρίας Φράγκα για να αναζητήσουμε μια λύση. Και τέλος επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελίας και όλους τους συζητητές για τη δουλειά τους. Ε, λυπάμαι που, ε, που μακρηγόρησα, αλλά είχα και εγώ τέσσερις εκθέσεις να σχολιάσω. Κυρία Επίτροπε, κυρία Δαμανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η Επιτροπή Προπολογισμών, ο συνάδελφος κύριος Αλφόνση, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό, ε, χρειάστηκε να εξετάσουμε την έκθεση αυτή για την αληφτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ένωσης των Κομόρων. Η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση αυτή, αλλά θεώρησε ότι ε, η ψήφιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χάνει το νόημά της από τη στιγμή που έγινε μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Και βεβαίως επειδή τα χρήματα είναι λίγα, ε, το, ο αντίκτυπος δεν είναι και τόσο σημαντικός. Καλό θα ήταν όμως να είχαμε την ευκαιρία να αποφανθούμε εξάντε. Από εκεί και πέρα αναλύσαμε ε, το θέμα σε βάθος, προστασία των αλευτικών πόρων από τη μία, αλευτική δραστηριότητα από την άλλη, ε, τοπι, ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη που να εφαρμόζεται σωστά από τη τρίτη. Όλα αυτά τα θέματα έχουν εξεταστεί και θα πρέπει η Επιτροπή για την Αλία να ε, ε για να εμβαθύνει σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ.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 Αξιότιμε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη ε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για άλλη μια φορά λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο πακέτο που αφορά στην αλληλευτική πολιτική. Εγώ ως συντονίστρια χαίρομαι που για τους δύο κανονισμούς βρήκαμε συμβαστική πρόταση με την ε, Επιτροπή και το Συμβούλιο για την έκθεση Γκρελιέ και για την έκθεση Φερέρα που αφορά το δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο. Όσον αφορά την Συμφωνία Λίας με τις Κομόρες και εκεί θα συμφωνήσουμε. Παρότι δεν θέλω να σας αποκρύψω ότι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ε, κοινή ελευτικής πολιτικής ε, θα ήθελα να υπάρχει μια τελείως διαφορετική εξέλιξη της Συμφωνίας Όμω, Όμως ε, προβλήματα υπάρχουν στη Ιρλανδία. Εκεί δεν γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητες ε, του Κοινοβουλίου και σιγά σιγά χάνω την υπομονή μου δεν έχουμε βρει ακόμα τη σωστή συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς και νομίζω αυτό το έχω πει επανειλημμένα και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Ε, το πρόβλημα των προγραμμάτων διαχείρισης πρέπει να λυθεί ταχύτατα και απευθύνω έκκληση στην Ουγγρική Προεδρία να ε, δραστηριοποιηθεί ε, για μία λύση. Το γεγονός ότι δεν έχουμε εδώ κανέναν από το Συμβούλιο αυτό καθιστά σαφές τον ελάχιστο σεβασμό ε, που δείχνει το Συμβούλιο προς το Κοινοβούλιο. Και άλλη μια παρατήρηση για την έκθεση Γκρεγέ. Γνωρίζω ότι ορισμένοι συνάδελφοι είναι απογοητευμένοι γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη οι τροπολογίες τους. Όμως είναι εξίσου κακό το ότι οι αλείς μας ε, είναι αναγκασμένοι να εργάζονται με πεπαλαιωμένα μέσα. Και εδώ φταίει το Συμβούλιο που δεν μπόρεσε να συμφωνήσει πάνω σε ένα καινούριο κανονισμό. Εμείς ε, ξέρουμε ότι ε, θα πρέπει να δράσουμε με υπευθυνότητα στο Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου ε, θα πρέπει τον υφιστάμενο κανονισμό να τον παρατείνουμε χωρίς αλλαγές. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος συνάδελφος, ο κ. Κέλαχα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τους τέσσερις εισηγητές για την παρουσίαση των εκθέσεών τους. Ε, έχετε τις παρατηρήσεις μου για την έκθεση Γκρέλια. Δεν θα μιλήσω πολύ για αυτή γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ως προς τα τεχνικά μέτρα. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στις ακτές της Ιρλανδίας και της Δυτικής Σκοτίας. Ε, κοιτάξτε, η μεταρρύθμιση κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, έχει δρομολογηθεί αλλά περιμένουμε και νέο κανονισμό. Καλό τις ε, πολιτικές ομάδες να στηρίξουν αυτές τις πολύ ρεαλιστικές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Τα μικρά αλλιευτικά σκάφη, μικρότερα των 15 μέτρων, δεν θα μπορούν να έχουν επαρκή εισοδήματα οι ιδιοκτήτες τους ενώ δραστηριοποιούνται σε πολύ επικίνδυνα νερά, καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Ουσιαστικά ε, κάνουμε αυτά τα σκάφη να πάνε μέσα μέχρι 80 χιλιόμετρα και παραπάνω για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τα δίχτυα που χρησιμοποιούν τα μικρά ε, αλλιευτικά σκάφη ε, για τα όστρακα δεν χρησιμοποιούνται για το γάδο ούτε ε, για άλλου είδους ίχθιες ε, που τα αποθέματά τους είναι εν κινδύνο. Επομένως, δεν αρκεί να πούμε ότι θέλουμε μόνο μία ανοιχτή συζήτηση. Τώρα, ως προς το βασιλάκι. Θα έλεγα ότι το Δεκέμβριο το Συμβούλιο ε, ε, θέτησε ε, συνολικό επιτροπόμενο αλίευμα συγκεκριμένο και στηρίχθηκε σε επιστημονικά δεδομένα. Όμως με τον υπάρχοντα κανονισμό δεν υπάρχει καμία αναφορά ως προς το είδος αυτό. Καλό να γίνει δεχτή η τροπολογία μου. Η πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιηθεί για να έχουμε ένα είδος, το μέγεθος του ματιού του δικτυού από 32 μέχρι 50. Και καλό τα κράτη-μέλη Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ακολουθεί η συνάδελφος κυρία Λούβιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, μέλη. Θέλω να συγχαρώ όλους τους ηγητές για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν και θα εστιαστώ στη συμφωνία με τις Κομόρες, με την Ένωση των Κομορών. Εμείς οι πράσινοι ψηφίσαμε όχι για αυτή τη συμφωνία και θα σας εξηγήσω γιατί. Η συμφωνία με τις Κομόρες που θα ψηφίσουμε αυτή είναι μια φτωχή χώρα με την οποία έχουμε συμφωνίες από το 88. Οι Κομόρες πήραν 2 εκατομμύρια ε, ε, ευρώ και ένα ποσοστό αυτών των χρημάτων προορίζεται για να έχει σκοπό να υποστηρίξει την τοπική αλία. Αυτή η αναπτυσσόμενη χώρα δεν έχει ούτε ένα, ένα λιμάνι που να λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν έχει καθόλου λιμενικό σώμα και ο τοπικός τομέας αλληλείας είναι πάρα πολύ πανάπτυκτος. 2,5 εκατομμύρια ευρώ παίρνουν οι κομόρες για τις και οι φορολογούμενοι πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού. Μιλάμε για αλία τόνου, για ε, τα σκάφη που προορίζονται για την αλία του τόνου, κατά κύριο λόγο. Οι, διοκτήτες, πλειοκτήτες είναι πολύ τυχεροί. Αλλά ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής ε, της συμφωνίας. Σε τι ωφελείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάρια δεν φτάνουν ποτέ στις Κομόρες, κανένας κάτοικος από τις Κομόρες δεν ε, εργάζεται σε αυτά τα πλοία. Το ερώτημά μου λοιπόν στην Επιτροπή είναι το εξής. Πώς θέλει, πώς πιστεύει θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα από την προηγούμενη αυτή η συμφωνία. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα, τα πλοία, θα, τα σκάφη θα χρησιμοποιούνται κάτοικοι των κομορών και πραγματικά θα βοηθηθεί θα βοηθηθεί η Ένωση των Κομορών από αυτή τη συμφωνία και δεν θα είναι απλώς αποφάσεις που θα μένουν στο χαρτί. Ευχαριστούμε την κυρία Λουβίν για 1,5 λεπτό. Ο συνάδελφος κύριος Γκρόμπατσικ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν ε, συντάσσοντας τις εκθέσεις τους. Οι εκθέσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές όσον αφορά στην κοινή ελευτική πολιτική. Βέβαια παράλληλα ε, πρέπει να ε, προβάλλουμε κάποια διάσταση απόψεων που υπάρχει ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες. Αν δούμε λιγάκι το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πούμε ότι η συνθήκη της ε, Λισαβόνας κατ' ουσίαν δίνει περισσότερες αρμοδιότητες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις ε, κανονιστικές διατάξεις και την σύναψη διεθνών συμφωνιών. Η Κομισιόν προσπαθεί να περιορίσει αυτές τις αρμοδιότητες όπως και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο κατ' ουσίαν πρέπει να έχει και ελεγκτικό, εποπτικό ρόλο οι ε, βουλευτές κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων πρέπει να μπορούν να κάνουν ακριβώς τη δουλειά τους. Η Επιτροπή ανταυτού ε, δεν θέλει να επιτρέψει στους βουλευτές να αναπτύσσουν αυτές τις ε, δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ περιορισμένες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για ένα λεπτό. Επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, μετά από ε, τόσα πολλά ε, χρόνια ε, υπήρξαν αλλαγές. Πριν από δύο χρόνια οι Σκοτσέζοι υπέβαλαν κάποιες, κάποια σχέδια αλλαγή και αυτό ήταν μια περιφερειακή προσέγγιση. Αλλά γιατί όχι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίζει, χωρίζεται σε περιφέρειες. Εμάς μας, ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρει το ότι πολλοί πηγαίνουν στις ε, Κομόρες ε, και λελατούν την περιοχή. Το ίδιο έχει γίνει και σε άλλες περιοχές. στη Σομαλία σας εκπλήσει το ότι εκεί εκεί κατέληξαν οι άνθρωποι στην πειρατεία. Ε, πριν από πέντε χρόνια είδαμε επίσης όλους αυτούς που ε, προσπάθησαν ε, να βρουν καταφύγιο στις Κανάριες νήσους. Μιλάμε ότι ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια όπου πάρα πολλοί πέθαναν πάνω στα αληφτικά σκάφη. Όμως δεν ενδιαφέρεστε για αυτούς τους ανθρώπους από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες γιατί αυτοί είναι πάρα πολύ φτωχοί, έχουν φτωχύνει περισσότερο περισσότερο από τις δικές σας τις πράξεις και γι' αυτό πρέπει να κατακρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κλακ. Η κυρία Ντότς για ένα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Ένας από τους εισηγητές μίλησε ε, για το ότι οι αλληλείς έχουν χάσει την πίστη τους στην αλληλευτική πολιτική. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει αυτό. Ουσιαστικά πιστεύουν ότι θα σημάνει την καταστροφή του στόλου τους χωρίς να έχουν ε, αυξηθεί και ε, διασφαλιστεί τα αποθέματα. Καλό θα ήταν η αλευτική πολιτική να επιστραφεί ως αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη. Το ταχύτερο δυνατό. Δυστυχώς όμως δεν θα γίνει αυτό, λίαν συντόμως. Και γι' αυτό έχω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχάς το θέμα της ε, δρέωσης ε, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει στα λευτικά πράγματα, ε, τουλάχιστον ας είναι σωστά χρηματοδοτούμενη η πολιτική της αυτή και να λαμβάνει υπόψη της η πολιτική ε, τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων. Οι αλλοί προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα κανόνων και κανονισμών, οι οποίοι θεσμοθετούνται χωρίς καν να ζητηθεί η γνώμη τους πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι στον τομέα αυτό, εμπλεκόμενοι στο κλάδο, μου έχουν μιλήσει και μου έχουν πει ότι ε, προσπαθούν αγωνιωδώς να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα πολύ περίπλοκα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ντότς. Ε, τώρα οι επόμενοι ομιλητές, ε, πρώτα απ' όλα ο συνάδελφος κύριος Καντέκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να σας μιλήσω από καρδιάς. Μία έδρα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Στρασβούργο. Θα ήθελα τώρα να συγχαρώ τον κύριο Φερέιρα για την έκθεσή του για τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την υλοποίηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής ε, και τα δικαιώματα ε, της θάλασσας ουσιαστικά. Μπορούμε να ε, χρηματοδοτήσουμε τις έρευνες και να συμβάλλουμε στη βελτίωση της κατάστασης μέσα στο πλαίσιο του κοινού νομοθετικού πλαισίου για τη συλλογή και χρήση όλων αυτών των στοιχείων και δεδομένων. Χαίρομαι ιδιαίτερος διότι ε, θα καταστεί δυνατό να χρηματοδοτηθεί η ερευνητική δραστηριότητα, η επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα για την αλία και την υδατοκαλλιέργεια. Ε, καλό θα ήταν να αναρωτηθούμε για το πόσο εξαρτώνται ε, οι εξαρτάται η ευρωπαϊκή αγορά από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Το ποσοστό είναι πάρα πολύ υψηλό και ε, όλο και αυξάνεται. Είναι απαραίτητο λοιπόν να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους παραγωγούς αν θέλετε και να μην ε, έχουμε άνοιγμα αγορών ε, εντάχει και χωρίς σωστή μέρημνα. Ε, ως προς την έκθεση Γκρελιέ, να συγχαρώ την εισηγήτρια. Τα τεχνικά μέτρα είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και θα πρέπει να λυθεί γρήγορα. Ε, να περιμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για τη δέσμη ε, που έχει να κάνει για το πακέτο μεταρρύθμισης της αλληλευτικής ε, πολιτικής. Θα ψηφίσουμε αύριο μια έκθεση η οποία θα, με την οποία θα δοθεί παράταση Άρα θα επιβιώσει ο κλάδος μετά τις 30 Ιουνίου αυτή της χρονιάς και θα ρυθμιστούν καλύτερα οι ελευτικές δραστηριότητες μέχρι ότου γίνει ε, πιο εις βάθος μελέτη ε, για τα τεχνικά μέτρα. Δεν είναι λογικό ε, να δεχθούμε επί της ουσίας τροποποιήσεις στην έκθεση αυτό στην έκθεση αυτή, γιατί αυτό συνεπάγεται μια επαχθή νομοθετική διαδικασία και ε, συζήτηση στο Συμβούλιο. Να συγχαρώ και τον κύριο Καπούλα Σάντο για τη διμερή συμφωνία με την Ένωση ε, της, για τι Κομόρε, αλλά και την συνάδελφο Φράγα για την έκθεση για την Γρυλανδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμεί για τα επόμενα δύο λεπτά. Συνάδελφο ε, Κρίστενσεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συζητητές ε, για το έργο τους. Αύριο λοιπόν ε, θα ψηφίσουμε για τη συμφωνία με τη Γρυλανδία και εγώ είμαι σκιώδης συγητής. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να απομακρύνουμε την ακριβή γραφειοκρατία και να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι κάτοικοι της Γρυλανδίας θα μπορούν να πολλούν τα προϊόντα τους εδώ στη δική μας ε, την κοινή αγορά εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές. Τα ψάρια της ε, Γρυλανδίας ε, σήμερα ελέγχονται καταρχήν στη Γρυλανδία και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτή τη συμφωνία θα πάψουν, να υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι. Αυτή λοιπόν η συμφωνία ε, θα φέρει μόνο ωφέλη. Και πέρασε πολύ καιρό να γίνει κάτι τέτοιο. Και είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο ε, προσέφερε τη νομική βάση και ελπίζω να την εγκρίνει το Συμβούλιο. Ε, εμείς συμφωνούμε αυτό αφορά αυτή τη συμφωνία με τις Κομόρες. Εμείς, εγώ είμαι υπέρ της ε, διάρκειας βιωσιμότητας ε, για τα λιεύματα, για το γηγενή πληθυσμό ε, και τέλος και βιωσιμότητα για όσου ε, χρησιμοποιούν αυτή τη συμφωνία. Όμω αυτή η συμφωνία με τι Κομόρε δεν είναι τόσο βιώσιμη όσο θα ήθελα γιατί δεν υπάρχει κανένα ανώτατο όριο για ε, τα αλλιεύματα, τα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Ε, όταν έχει συμπληρωθεί το απαραίτητο ποσό, μετά για κάθε τόνο καταβάλλονται 65 μόνο ευρώ. Η τάση λοιπόν θα πρέπει να είναι να υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο αυτό είναι επιζήμιο και λάθο. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε ε, μία ε, λανθασμένη πολιτική ε, στα δικά μας αλλά ούτε και στα ξένα είδατε. Εγώ θέλω τα χρήματα που καταβάλλονται ως αντιπαροχή για αυτές τις συμφωνίες της Αλίας να χρησιμοποιούνται για το γηγενή πληθυσμό. Σε αυτούς να φτάνουν τα χρήματα. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε, κύριε Κρίστενσεν για ένα λεπτό η συνάδελφος κυρία Ράιμερς. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Ανταμανάκη, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που επιτέλους ε, το θέμα αυτό ε, θα ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τους εισηγητές για την εργασία τους. Η τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική. Και αυτό ισχύει κυρίως για τους τομείς διεθνής αλληλευτικές σχέσεις, συγκέντρωση δεδομένων και επιστημονικές μελέτες. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ελεγκτικά συστήματα της κοινή ελεγκτικής πολιτικής. Ο εισηγητής προσπάθησε ε, να πείσει τους συναντέλφους του γιατί ε, πρέπει να φτάσουμε ε, το όριο στο 65%. 75% με Ο κανονισμός αποδείχτηκε σωστός στην πράξη. Τα κράτη-μέλη ε, ήδη τώρα καταφεύγουν στη δυνατότητα της ε, συγχρηματοδότησης και δεν χρειάζονται περαιτέρω κίνητρα. Είναι λοιπόν σημαντικό με την τροποποίηση του κανονισμού να ανοίξει ο δρόμος για ένα ε, συνεπή, συνεπές νομικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε, λέει ο για ένα λεπτό συνάδελφος Χάτσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση Γκρελιέ παραχωρεί υπερβολικά πράγματα στην Επιτροπή οι αλληλείς της Σκοτίας δυσκολεύονται να καταλάβουν γιατί η Επιτροπή καταργεί ορισμένα πράγματα ενώ ε, δεν δέχεται τις ε, ορισμένες ε, τροπολογίες. γιατί η παράταση για ακόμα 18 μήνες προσωρινών μέτρων όπως τα ονομάζει η Επιτροπή για την προστασία των αποθεμάτων. Καλό τους συναδέλφους αύριο να υποστηρίξουν όλες τις τροποποίησεις στη διάρκεια της ψηφοφορία και ελπίζω ότι οι τροποπλογίες θα εγκριθούν και αν εγκριθούν ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αλλάξει στάση και θα αδράξει την ευκαιρία που της προσφέρεται να ενεργήσει με διαφορετικό τρόπο και όχι τώρα άμεσα και όχι κάποτε στο μέλλον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχω υποβάλει τροπολογία ε, ως προς την έκθεση των τεχνικών ε, μέτρων για να ε, λυθεί το θέμα που έχει να κάνει με τις δυτικές ακτές της Σκοτίας, ώστε να διατηρηθούν τα αποθέματα ηχθείων λευκής σαρκός. Ε, για 12 μήνες είχαν θεσπιστεί αυτοί οι προσωρινοί κανόνες, δόθηκε παράταση βάσει της συμφωνίας Catch All και ε, τώρα η Επιτροπή θέλει να ξανα καμψει αν θέλετε τους κανόνες και να πάμε μέχρι το 2012 μέχρι να καταρτιστεί νέο πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα βάσει της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Άρα ένας προσωρινός κανονισμός που ουσιαστικά υιοθετήθηκε μόνο για ένα χρόνο θα εφαρμοστεί για τρία χρόνια, μία περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες στις δυτικές ακτές της Σκοτίας έχουν αλλάξει ε, τα μάλα, αναγκάζοντας ε, τους ε, αλληλείς μας να απορρίπτουν αλλιεύματα πολύ σημαντικά ε, στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά, επόμενος ομιλητής, Πατράωνεβες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές και θα σε δύο εκθέσεις. Το 2008 με βάση ένα σχέδιο κανονισμού που θα έχει σκοπό να πλουστεύσει ένα κοινοτικό κανονισμό που αφορούσε τη συντήρηση, τη διατήρηση των αλλιευτικών πόρων, οδήγησε στην ψήφιση του σημερινού κανονισμού που προβλέπει μια σειρά από μεταβατικών μέτρων που είχαν αρχικά προβλεφθεί για μια περίοδο μεταξύ 1η Ιανουαρίου 2010 και 30 Ιουνίου 2011 η σήμερα θα παραταθεί αυτό το μεταβατικό καθεστώς επί 18 μήνες, δηλαδή μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2013. Στο μεταξύ, περιμένοντας ένα νέο κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα που θα πλαισιώσει τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής πρέπει να διατηρήσουμε ένα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Ελία, να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των αλλιέων, χωρίς να χάσουμε ε, το σημαντικό στόχο που είναι η δημιουργία μιας αηφόρου Ελίας. Η μη ε, παράταση σε ό,τι η, χρήση ε, συγκεκριμένων δικτυών χωρίς να υπάρχουν ε, βάσιμα ε, επιστημονικά στοιχεία δεν είναι κάτι το σωστό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι βιοτέχνες αλληλείς της ε, Πορτογαλίας χρησιμοποιούσαν αυτά τα δίχτυα και η κατάργησή τους είναι ένα πλήγμα για την κοινότητα των αλλιέων που εξαρτάται για την επιβίωσή της από την αλλία. Θα ήθελα λοιπόν να εγκριθεί μια πρόταση που ε, υπέβαλαν ο συνάδελφος Κάπουλα Σάντος και άλλοι μαζί μου ώστε να διατηρηθεί για διατηρηθεί με το 2013 μια κατάσταση που δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τους αλείς. Τώρα, για το, δικαίωμα, για το δίκαιο ε, της θάλασσας και την μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής. Το Ταμείο Λύσης είναι το σημαντικότερο μέσο που επιτρέπει τη χρηματοδότηση ε, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης δεδομένων, της επιθεωρήσης, τους ελέγχους για την εφαρμογή της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Επ' αυτού συμφώνησα απόλυτα με την πρόταση του εισηγητή στην Ολομέλεια που, που, προέβλεπε την αύξηση του, της κοινοτικής χρηματοδότησης μέχρι του 60% σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση θεμελιωδών δεδομένων και την συγκέντρωση και τη διαχείριση πληρωματικών στοιχείων. Η ευρύτερη γνώση και η γενική ευμένη γνώση ε, τη, των συνθήκων αλίας και η ανάγκη η αλία να στηρίζεται πάνω σε επιστημονικά δεδομένα είναι κάτι το πολύ σημαντικό και γι' αυτό υποστηρίζουμε την έκθεση. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος ε, Ανδρέας Μπαρέα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους τέσσερις εισηγητές για την εξαιρετική τους εργασία. Ε, δεδομένη της σημασία που έχουν οι εκθέσεις ε, αυτές, θα ήθελα καταρχάς να σχολιάσω ε, τη συμφωνία με τις Κομόρες Νήσους. Έχουμε μια νέα συμφωνία με μια χώρα που βρίσκεται ουσιαστικά στην, κοντά στην Νοτιοανατολική Αφρική, και το 60% του πληθυσμού διαβεί κάτω από το κατόφλι, το όριο της φτώχειας. Και ο μόνος τρόπος επιβίωσης είναι να αυξηθεί ο τουρισμός ή να έχουν πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις. Ε, είναι η δυνατότητα να αλλιεύουν το, την, τα υπερβάλλοντα, τα πλεονασματικά αλλιευτικά ε, αποθέματα. Και το λέω ε, ε, διότι έτσι βοηθείται η χώρα αυτή να βελτιώσει τις υποδομές της για να αυξήσει την, ε, και να προσελκύσει τουρισμού και να αναπτυχθεί καλύτερα. Μιλούμε για μια βιώσιμη υπεύθυνη αλληλεία διατηρώντας τους θαλασσιούς πόρους. Μεταναστευτικά είδη όπως τα τονοειδή περνούν από την περιοχή αυτή και κάθε χρονιά καθορίζεται το απόθεμα για την επόμενη χρονιά βάσει επιστημονικών μελετών και επί την παρουσία συγκεκριμένων παρατηρητών. Ε, μιλάμε για την παράκτη αλία στην ε, περιοχή αυτή ώστε ε, να είναι βιώσιμη. Το πρωτόκολλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι τα αλλιευτικά σκάφη τα ευρωπαϊκά θα έχουν πρόσβαση στην περιοχή αυτή και θα βελτιωθούν και οι οικονομικές προοπτικές. Η συμφωνία έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία διότι έτσι δεν γίνεται αλία, από τρίτες χώρες οι οποίες δεν έχουν τόσο υψηλά στάνταρ περιβαλλοντικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό το αλλιεύεται από τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι είναι μια συμφωνία που βοηθάει ιδιαίτερο στις κομμόρες νήσους αλλά προστατεύει και το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σχολιάσω επίσης και την έκθεση της κυρίας Γκρελιέ για τα τεχνικά μέτρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ε, ζητείτε παράταση μέχρι το Δεκέμβριο του 2012. Αλλιώς θα υποπέσουμε σε νομικό κενό και θα υπάρξει νομική ασάφεια και κακή βεβαίως διατήρηση των θαλάσσιων πόρων. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία η δήλωση, η συνημένη δήλωση. Ζητείτε από την Επιτροπή να δεχθεί συγκεκριμένες τροποποιήσεις στα τεχνικά μέτρα έτσι όπως τα έχουν προτείνει ορισμένα κράτη-μέλη. Μιλούμε για το μάτι ε, του δικτυού αλλά και το βάθος. Σε τι βάθος γίνεται αλληλεία, ε, αλληλευτική δραστηριότητα. Θα πρέπει η Επιτροπή να τα λάβει υπόψη της αυτά, να δει ε, πόσο θα επηρεαστούν τα αποθέματα στις ζώνες 8, 9 και 10 Ουσιαστικά πρόκειται για ελλείψεις, για κενά στην εφαρμογή του κανονισμού που ε, πλήττουν την αλληλευτική δραστηριότητα αλλά και τα αποθέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπιλμπάο Μπαράντικα, η συνάδελφη κ. Μπιλμπάο Μπαράντικα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα υπερψηφίσω την έκθεση αυτή γιατί θα ευνοήσει τον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο 70 σκάφη ε, και θα υπάρχει και ένα μέλος του πληρώματος το οποίο να προέρχεται από τις νήσους Κομόρες. Άρα προστατεύονται και οι θέσεις απασχόλησης εκεί. Είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται σε διμερή συνεργασία, αναπτύσσεται η περιοχή. Καλή αμφότερα μέρη να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι, η σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στοιχείο κλειδί για να συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία. Στηρίζονται οι παραδοσιακές τεχνικές αν θέλετε, αλλιευτικέ πρακτικές. Και αυτές οι λίγες χιλιάδες άνθρωποι από τι νήσε Κομόρες θα έχουν ε, δικά του αλλιευτικά σκάφη, θα μπορέσουν να συνεχίσουν την αλλιευτική του δραστηριότητα. Προωθεί η συμφωνία αυτή ε, την βιωσιμότητα της αλίας στην περιοχή και υπάρχουν και μηχανισμοί για την επιστημονική συνεργασία και την καλύτερη εξαγωγή των πορισμάτων. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος κύριος Κέλλη. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ομιλώ εξ ονόματος της ομάδας μου για αυτό το θέμα που είναι ομολογώ ιδιαίτερα επίμαχο ένα από τα πιο επίμαχα που χρειάστηκε να συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οφείλεται στο, στους αλληλείς και στην αλληλεία που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι δυνατό να μιλήσουμε για όλα τα τεχνικά θέματα, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Μας παρουσίασε μια εικόνα της κατάστασης η Επίτροπος υπάρχει θέμα αρμοδιοτήτων έναντι του, του Συμβουλίου αλλά όπως είπατε θα βρεθεί κάτι και αυτό είναι επιθυμητό μια ρεαλιστική λύση αλλά ίσως πιο σημαντικό είναι να βρεθούν λύσεις για χώρες που εξαρτώνται από την αλία για την επιβίωσή της και για την ανάπτυξη της οικονομίας της. Για τη συμφωνία μπορούμε να πούμε ότι τα ψάρια που θα προέρχονται από αυτή την περιοχή θα είναι ύψης της ποιότητας και θα έχουν ελεγχθεί σωστά διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα, τις τεράστιες υδατοκαλλιέργειες στην Νοτιοανατολική Ασία. Ε, καλούμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε σημαντικότατα θέματα όπως είπε και σήμερα το απόγευμα η Επίτροπος, η κατάσταση σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των κοινοτήτων και των αλλιευτικών πόρων ε, αμφισβητείται. Χρειάζονται λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη στα πλαίσια της αναθεώρησης της κοινή ελευτικής πολιτικής. Αλλά εντωμεταξύ δέχομαι την έκθεση, μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση και συμφωνώ με αυτά που μας είπε η Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Κέλλη. Σάντσες Πρεσέντο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ με τη σειρά μου τους τέσσερις εισηγητές και θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου ε, στην έκθεση ε, Καπούλας Σάντος ως προς την ε, χρηματική αντιπαροχή και τη συναλλευτική δραστηριότητα με τις, που όπως εκφράζονται συμφωνία με τις νήσους Κομόρες. Συμφωνώ και με την ουσία της έκθεσης της κυρίας Γκαλιέ για τα τεχνικά μέτρα. Θα πρέπει η Επιτροπή να επιταχύνει την αξιολόγηση του αντικτύπου ώστε να έχουμε ένα νέο κανονισμό για αυτά τα τεχνικά μέτρα και να υιοθετηθεί αυτός ο κανονισμός το ταχύτερο δυνατό και ή δυνατό πριν από το 2013. Η έκθεση Φορέιρα τροποποιεί το κανονισμό 812 ε, ε, του 2006 ε, λαμβάνοντας υπόψη τα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση που αναλογεί στη κοινή αλληλευτική πολιτική ε, με την καινούργια συνθήκη. Είναι μια έκθεση την οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Είναι σημαντική η βιώσιμη και να για να υπάρξει η βιώσιμη θα πρέπει να υπάρχει και βιώσιμη αλληλευτική δραστηριότητα αλλά και ε, προστασία των αποθεμάτων. Ε, μπορέσαμε έτσι να αυξήσουμε τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Η έκθεση Φράγα έχει να κάνει με ε, την τήρηση υγειονομικών πρακτικών και κανόνων έτσι ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή ε, αλλιευτικών προϊόντων και υποπροϊόντων από την Γρυλανδία. Οι κανόνες αυτοί αφορούν το 90% των εξαγωγών της Γρυλανδίας. Το 2007 οι εξαγωγές αυτές έφτασαν, ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσει η Γρυλανδία τα, αυτά που ισχύουν στην εσωτερική αγορά. Έτσι θα διευρύνουμε την ενιαία αγορά. Προφανώς. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για τη νομική βάση και γι' αυτό θεωρώ ότι η Επιτροπή έχει πολύ καλή στάση, διότι η Επιτροπή ενθαρρύνει την επίτευξη συμφωνίας. και καλό θα είναι να ληφθεί υπόψη η θέση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων που στηρίζει την άποψη της Επιτροπής Αλίας. Η Γρυλανδία είναι ένα θέμα υψηλής προτεραιότητας και ελπίζουμε να λυθεί σύντομα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Για ένα λεπτό η συνάδελφος κυρία Ντάνκυλα. Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ και τους τέσσερις εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν για τον τομέα της αλίας και να υπογραμμίσω ότι τα χρηματοδοτικά ε, μέσα για την εφαρμογή της ενιαίας κοινή αλλιευτικής πολιτικής σημαίνει μια τεράστια χρηματοδότηση της αλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέτρα αυτά πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πολιτών λαμβάνοντας υπόψη και τις σημερινές προκλήσεις. Τα χρηματοδοτικά, τα οικονομικά μέσα για την εφαρμογή της ε, κοινή αλλιευτικής πολιτικής περιλαμβάνουν έργα όπως το τομέα των δημοσίων σχέσεων, των διεθνών σχέσεων, τη συγκέντρωση στοιχείων, την επιστημονική ανάλυση, τη διακυβέρνηση και την εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η διαχείριση της αλληλείας πρέπει να στηρίζεται σε ε, σύγχρονα ε, επιστημονικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την κατάσταση των αλλιευτικών πόρων και με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Τάνκυλα. Ε, δεν ε, έχει πλέον κανείς άλλος ζητήσει το λόγο. Περνάμε... Κανείς δεν έχει ζητήσει το catch the eye το λόγο και γι' αυτό δίνω κατευθείαν το λόγο στην κυρία Δαμανάκη. Θα ήθελα να σας ε, δώσω κάποιες σύντομες εξηγήσει μετά από τις παρατηρήσεις σας. Αναφερόμενοι στη συζήτηση και στην εταιρεία σύμπραξης για την Αλία θα σας πω ότι στα πλαίσια της πρότασής μας θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των συμφωνιών αλίας ώστε να αποβούν προς όφελος για τον τοπικό πληθυσμό. Έως ότου έχουμε τις νέες προτάσεις για τη νέα γενιά αλλιευτικών συμφωνιών θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την σημερινή κατάσταση και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα καταβάλουμε προσπάθεια, κάθε προσπάθεια, ώστε να υπάρξει καλή, σωστή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με τις Κομόρες, προς όφελος, όπως είπα προηγουμένως, του τοπικού πληθυσμού. Τώρα, σχετικά με τα προβλήματα που αναφέρθηκαν ε, σε σχέση με το Κοινοβούλιο και την ενημέρωση των μελών του Κοινοβουλίου για τις διάφορες συμφωνίες μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει ε, όλες, ακόμα όλες τις, ε, τις πληροφορίες και όλα τα κείμενα των συμφωνιών στο Κοινοβούλιο, ακόμα και τις, συμφωνί, τις, τα στοιχεία που είναι απόρριτα και αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ανησυχίες για την παράταση του κανονισμού του ισχύοντος κανονισμού, χρειάστηκε να το κάνουμε αυτό, διότι έπρεπε να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταρρύθμισης αλλά αντιλαμβάνομαι γιατί μας καλείται να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να έχουμε ένα νέο κανονισμό πριν από το τέλος του 2013. Δεν μπορώ να σας δώσω υποσχέσεις που δεν, είμαι βέβαιη να τηρήσω, ότι θα τηρήσω, αλλά σας λέω ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να επιταχύνουμε τη διαδικασία για, για ένα νέο κανονισμό και για την εφαρμογή του βασικού κανονισμού για τη μεταρρύθμιση ώστε να αναλάβουν κάποιες αρμοδιότητες σχετικά με τα τεχνικά μέτρα τα κράτη-μέλη. Το επόμενο θέμα, ο δημοσιονομικός κανονισμός, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια πρώτη ανάγνωση, θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση της ε, ε, πρώτης ανάγνωσης. Και για τη Γρυλανδία τέλος, επαναλαμβάνω και πάλι ότι αναζητούμε λύση για την νομική βάση της πρότασης για την Επιτροπή. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να προχωρήσουμε διότι η Γρυλανδία και οι καλές σχέσεις με τη Γρυλανδία αποτελούν απόλυτη πολιτική προτεραιότητα για μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η Επιτροπή είναι εδώ για να διευκολύνει και να αναζητήσει μια συμβιβαστική λύση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, κυρία Δαμανάκη. Οι εισηγητές θα συνοψίσουν ε, τις παρεμβάσεις τους. Ο κύριος Καπουλασάντος θα είναι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, σας ευχαριστώ για αυτά, για, για όσα ελέγχθησαν για το άτομό μου. Και οπωσδήποτε απαντήθηκαν ορισμένα ε, από τις προσδοκίες και τα ερωτήματά μου. Αυτές οι ε, συμφωνίες σύμπραξης πρέπει να μελετηθούν ε, ε, δέχομαι, δέχομαι ε, τη θέση της, της Επιτρόπου σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των Ευρωβουλευτών και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ταχύτερα η εκπλήρωση και η υλοποίηση των στόχων μας. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Φερέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές για όλα τους τα σχόλια. Είναι πολύ ε, σημαντικό το θέμα και όλοι ενδιαφέρονται να προχωρήσει προς τα εμπρός. Ως προς τα ε, χρηματοδοτικά μέτρα και τις προτάσεις μας, θα ήθελα να πω ότι, το, ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα συνένεση. Ελπίζω να υπάρξει λίαν συντόμως συνένεση. Πολλοί συνάδελφοι στήριξαν τις προτάσεις αυτές και χαίρομαι γι' αυτό. Η βάση για την έγκριση της, ε, των τροπολογιών αυτών θα ήταν κάτι το πολύ θετικό. Από τη μία η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή. Από την άλλη όμως ουσιαστικά ε, είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Τώρα, ως προς την έκθεση για ε, τα μεταβατικά μέτρα, θα ήθελα να τονίσω ότι η τροπολογία που έχω αποβάλει εγώ μαζί με άλλους δύο συναθέλφους για να μην υπάρχουν πλέον αρνητικές διακρίσεις ε, βασίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επιστημονικό θεμέλιο, επιστημονική βάση που να ε, δικαιολογεί αυτές τις αρνητικές διακρίσεις. Η στόλη, η αυτοί αυτή στόλη, δείχνουν ότι χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα αποθέματα ε, στη γλώσσα για παράδειγμα, αλλά και σε άλλα είδη. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να στηρίζουν την άποψη αυτή και η απουσία επιστημονικών στοιχείων ουσιαστικά ενισχύει τη δική μας τη θέση να σας πω ότι στηρίζουμε τις προτάσεις των Ιρλανδών και Σκοτσέζων συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία, κύριε Φερέρα. Η κυρία Γκρελιέ. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε να μιλήσω πιο αργά αυτή τη φορά. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους που υποστηρίζουν την έκθεση μετά από τη συζήτηση που είχαμε στη διάρκεια της, στις Επιτροπή Ελίας. Συμμερίζομαι την άποψη της ε, ε, Επιτρόπου σε ό,τι αφορά το μέγεθος του ματιού για το βασιλάκι και ότι δεν πρέπει να αλλάξουν ορισμένα τεχνικά μέτρα που δεν υποστηρίζονται εφόσον αυτά τα επιστημονικά δεδομένα δεν έχουν διαβιβαστεί από τα κράτη-μέλη και επειδή όλα τα μέτρα που συνδέονται μεταξύ τους δεν έχουν όλα αξιολογηθεί. Επιμένω, όπως το έκαναν και οι προηγούμενοι ομιλητέ για το γεγονός ότι επήγει για η Επιτροπή να προβεί στην αξιολόγηση των ε, μέτρων αυτών και να προτείνει μια νέα, και να προ, προτείνει μια νέα πρόταση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ε, κοινής ελληνευτική πολιτική και όχι μετά την ολοκλήρωση. Τη τη βούληση που εκφράσατε να επιταχύνετε τη διαδικασία της πρόταση, κυρία Επίτροπε και ολοκληρώνοντας θυμίζω τη σημασία της κοινή προσπάθειας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, λιευτικών οργανώσεων για κάτι που θεωρώ σαν ε, απαραίτητο για μια υγιή αλία που θα διαθέτει τα αναγκαία μέσα που εξασφαλίζουν ε, έτσι ε, την επιβίωση και την ε, συνέχιση της δραστηριότητας όλων των ενδιαφερομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχα... Κυρία Γκρελιέ, η κυρία Φράγα, πρόεδρος της Επιτροπής Αλίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Επίτροπο γιατί απάντησε πολύ καλά στην ε, ερώτησή μου και είπε ότι ε, διατίθεται να δεχθεί την τροποποίηση της νομικής βάσης και ελπίζω και το Συμβούλιο να ακολουθήσει τη γραμμή της αξιότιμης κυρίας Επιτρόπου. Σε κάθε περίπτωση σκέφτηκα κατά πόσο είναι εφικτό αύριο να ζητήσω να ξαναπάει το θέμα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πριν ψηφιστεί οριστικά. Στη με συνέχεια σκέφτηκα ότι αν ζητήσω κάτι τέτοιο το μόνο που θα πετύχω είναι να καθυστερήσει η έγκριση ενός θέματος το οποίο ουσιαστικά ωφελεί και την Γροϊλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα είναι λοιπόν να μην το καθυστερήσουμε. Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ε, το Συμβούλιο να κινηθεί τάχιστα και να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα της δικής μας Επιτροπής. Ε, διότι επαναλαμβάνω το θέμα έχει να κάνει με την νομική βάση ενώ επί του περιεχομένου είμαστε όλοι σύμφωνοι. Χαίρομαι που ολοκληρώσαμε την εξέταση όλων αυτών των θεμάτων. Πάντοτε υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εμείς θα δείξουμε καλή θέληση αύριο και ελπίζουμε το Συμβούλιο να ανταποκριθεί όπως πρέπει. Επαναλαμβάνω για εμάς, αύριο είναι πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ και πάλι την ε, κυρία Επίτροπο για την πολύ καλή της συνεργασία. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου και που εκφράζουν τη στήριξή τους στην έκθεση αυτή. Επαναλαμβάνω, το μόνο που ελπίζουμε είναι το Συμβούλιο να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματά μας τα οποία στηρίζει και η Επιτροπή Νομικών Θωμάτων αλλά και η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία ε, Φράγα Εστέβεθ. Ε, ολοκληρώνεται η συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Ψηφοφορία λοιπόν αύριο στις 12. Αύριο Τετάρτη 6 Απριλίου συνεχίζεται η Ολομέλεια από τις 9 μέχρι τη 1, από τις 3 μέχρι τις 8. Θα σας μοιραστεί η μερίσια διάταξη, η οποία βρίσκεται